Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, καθίστε. Σας ε, καλωσορίζω μετά την εντατική προηγούμενη εβδομάδα συνεδριάζουμε ξανά σήμερα. Πρώτα απ' όλα, η μερίσια διάταξη την έχετε λάβει. Θέλετε να αλλάξει τίποτα. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να αναφέρω το γλωσσικό καθεστώς. Να πω πως το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασης μας θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο και οποιοδήποτε ε, λάβει το λόγο αυτομάτως θα φαίνεται κιόλας. Μετά, τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε τελειώσαμε και με αυτό το σημείο και θεωρούμε πως έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Περνάμε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 4. Ο ορισμός δύο μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και ακρόαση των υποψηφίων. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία υποψήφιο την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα από την Βουλγαρία. Η δεύτερη ε, ακρόαση ε, που αφορούσε την υποψηφία από τη Ρουμανία αναβλήθηκε γιατί μας είπαν ε, πως η υποψηφιότητα του Μυρσέα Βασίλε Ποπέσκου αποσύρεται Οπότε δεν θα έχουμε σήμερα την ακρόαση του κυρίου Ποπέσκου. 31 Δεκάτου βεβαίως αυτού του έτους ε, λίγη η θητεία των μέλων του ελεγκτικού συνεδρίου και θα πρέπει άρα να αντικατασταθούν τα μέλη αυτά και σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 της συνθήκης ε, το Συμβούλιο μετά από την διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει τη σχετική απόφαση γι' αυτό σήμερα έχουμε την ακρόαση της ε, υποψηφίας που προτείνεται από τις βουλγαρικές αρχές της κυρίας Ιβάνοβα. Έχουμε βεβαίως ε, μοιράσει και το ερωτηματολόγιο για να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι υποψήφοι, οπότε αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ακρόαση. Η ακρόαση θα λάβει χώρα τώρα. Θα ήθελα να προσκαλέσω την υποψήφια να κάνει μια αρχική τοποθέτηση 5 λεπτών και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ερωτήσεις ε, στην υποψήφια. Μετά δε το δημοσιότημα της ε, συνεδρίασης ε, θα περάσουμε και σε ένα κομμάτι που θα είναι και κλεισμένων των θυρών και θα αφορά την αξιολόγηση. οπότε μπορούμε να περάσουμε απευθείας στη συνέχεια της διαδικασίας. Κύριε Ιβάνοβα, σας ε, καλωσορίζω. Δεν χρειάζεται συστάσεις ε, στην Επιτροπή μας. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Τόλερ, αγαπητή κυρία Γιάλα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι χαρά και τιμή για μένα να είμαι μπροστά σας σαν υποψήφια από τη Βουλγαρία για μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Θεωρώ ότι είναι προνόμιο αυτή η υποψηφιότητα αλλά και τεράστια ευθύνη που αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενα σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνέδρου όσον αφορά τη διαδικασία του προπολογισμού, κυρίω στο παρόν οικονομικό περιβάλλον στην παρουσίασή μου σήμερα θα προσπαθήσω για περίπου ένα πεντάλεπτο να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ελπίζω θα σας βοηθήσουν να πάρετε μια ξεκάθαρη απόφαση μετά την ακρόαση. Και αυτό το ερώτημα είναι ποιος είμαι εγώ, τι έχω κάνει στην επαγγελματική μου ζωή και γιατί θέλω αυτή τη θέση. Για να σας ενημερώσω για να μπορείτε να κρίνετε γιατί αξίζει τη εμπιστοσύνη σα, Όπως θα βλέπετε από τι απαντήσεις των γραπτών ερωτηματολογίων που σας έδωσα, έχω 12 χρόνια συνολικά επαγγελματικής και πολιτικής εμπειρίας σε διάφορες κυβερνήσεις, σε πολιτικούς και ιδιωτικού φορείς. Έχω δύο πτυχία μάστερ σε διεθνεί οικονομικέ σχέσει και διεθνή διαχείριση και χρηματοπιστωτικά θέματα ε, από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές των θέσεων που κατήχα που θεωρώ ότι ε, ταιριάζουν πολύ με το ρόλο ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνέδριου. Πρώτα απ' όλα η εμπειρία μου όσον αφορά το κυβερνητικό τομέα στην Βουλγαρία σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο όταν ήμουν συντονίστρια για διεθνή χρηματοστατικά ιδρύματα στο Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων. Ε, Εντό των πλαισίων αυτών των ευθυνών συμμετείχα σε ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα ύψου 50 εκατομμυρίων Αμερικανικών δολαρίων για τη μεταρρύθμιση τη βουλγαρική γεωργία, ώστε να δημιουργήσουμε διοικητικό δυναμικό και να προετοιμάσουμε τον τομέα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό τμήμα τη εργασία μου τότε σχετιζόταν στον εκτοριστέρων έλεγχο των προγραμμάτων, όπου ήμουν υπεύθυνη για την αξιολόγηση ε, της γενικής αποτελεσματικότητας ε, εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων. Η εμπειρία που είχα στο Υπουργείο πριν το 1999 μου θυμίζει κάποια από τα μέτρα και μεταρρυθμίσεις που κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν τώρα, κυρίως με την εφαρμογή του νέου μακροχρηματοστικού μέσου, των νέων μέσων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης, παρόμοια στο ζύγια πληρωμών παρόμοιος τρόπος ελέγχου μέσω ε, μητρών ε, μετρήσεων και πιστεύω ότι η εμπειρία μου ε, όσον αφορά αυτά τα θέματα θα είναι κάτι πολύτιμο το ελεκτικό συνέδριο για περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας ελέγχου του προπολογισμού όσον αφορά τα ανέγνωτιστικά μέσα. Παρόμοια σημαντική εμπειρία μου και είναι ιδιωτική εμπειρία όταν δούλευσα σε τράπεζες και χρηματοστικά ιδρύματα στον τομέα του ελέγχου ε, των χρηματοδοτικών αυτών φορέων στη ΣΥΠΑ. Η εμπειρία μου όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου ήταν κάτι που βοηθά πολύ, κυρίω για να μπορέσω να καταλάβω εκ των κάτω προ τα πάνω την δημοσιονομική διαχείριση. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, να αναφέρω κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκα εδώ, επικοδομητικά, συνεργαζόμενοι με πολλού από εσά στην Κοκομπού, όπω είναι νετήσια έκθεση του 2010 ε, τι νομοδοτήσει για τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στα πλαίσια του νέου πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου, ε, την κοινή αγροτική πολιτική, το θέμα για το Hercule 3, πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την προστασία των χρηματοπιστωτικών συμφερόντων τη Ενώσεω, η μελέτη όσον αφορά το ESM και το FSM και πώ υπάρχει αλληλεπίδραση όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου του προπολογισμού και ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλο κάτι εξίσου σημαντικό Ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου του 2010 και για την απαλλαγή του 2009 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτό το ιστορικό δίνουμε την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, γιατί θέλω αυτή τη θέση. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποια είναι η απάντηση, όχι μόνο διότι θεωρώ ότι έχω αποκτήσει την αναγκαίε ικανότητε και δεξιότητε γι' αυτό. Επίση όμω, διότι ενδιαφέρομαι πολύ για θέματα ελέγχου του προπολογισμού και νομίζω ότι έχω αποδείξει με τη δουλειά που έχω κάνει μέχρι τώρα ότι είμαι αφοσιωμένη στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι η συνεχισή και εμβάθυνση αυτού του είδους του έργου στο ελεκτικό συνέδριο είναι κάτι μόνο φυσικό. Θα δώσω προστιθέμενη αξία όχι μόνο στα μέλη αυτής της Επιτροπής αλλά και για τις συζητήσεις που συνεχίζονται στο Λουξεμβούργο και αφορούν τις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το ελεκτικό συνέδριο. Κάποιες από τις ερωτήσεις νομίζω ότι θα μπορούσα διάφορα θέματα θα μπορούσα να βοηθήσω είναι τα χρηματοδοτικά μέσα, να δώσω προστιθέμενη αξία σε αυτό το τομέα. Και ένα από τα πιο ισχυρά μου σημεία σχετίζεται με τους ελέγχους επιδόσεων και τις ειδικέ εκθέσεις που εκπονεί το ελεγκτικό συνέδριο και θα προσπαθήσω τόσο σε αυτές οι εκθέσεις ε, να έρχονται πιο έγκαιρα, να είναι πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερε ανάγκες των μελών της Επιτροπής αυτής. Εάν ε, με υποστηρίξετε και εγκρίνετε την ε, διορισμό μου, θα συνεργαστώ μαζί σας μέσω συνεχούς διαλόγου και συνεργασίας και μαζί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Äh, σας ευχαριστώ κυρία Ιβάνοβα για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις σας. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Πρώτα, αν θέλει, θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία εισηγητριά μας, στην κυρία Αγία Σέμπερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω την κυρία Ιβάνοβα. Είδαμε πρόσφατα τη γαλλική κυβέρνηση και τους διορισμούς που κάνουν άλλες κυβερνήσεις ε, για το Ελεκτικό Συνέδριο με συναδέρφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δίνει μια μεγάλη προβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι σημαντική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ίσως δεξαμενή για στελέχωση σημαντικών ε, άλλων θεσμικών οργάνων. Είναι σημαντικό λοιπόν που μας παρουσιάσατε και το βιογραφικό σας και κάποια στοιχεία της πολιτικής και επαγγελματικής σας πείρας. Συμμετείχατε άλλωστε και σε προηγούμενες ακροάσεις και έχετε πλούσια πείρα από τα θέματα αυτά. Μας μιλήσατε εδώ για την 12 η σας πείρα. Μας εξηγήσατε διεξοδικά σε τι έγκυται αυτή η επαγγελματική και πολιτική πείρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στο ελεκτικό συνέδριο της Βουλγαρίας απαιτείται 15 ετή πείρα για να μπορεί κανείς να υποβάλει την υποψηφιότητά του για το βουλγαρικό ελεκτικό συνέδριο. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι με 12 μόνο χρόνια πείρας όπως προκύπτει από το βιογραφικό σας και δεδομένου του νερού τη ηλικία σας. Πιστεύετε ότι με αυτή την πείρα είστε έτοιμοι, είστε προετοιμασμένοι για να αναλάβετε τη θέση σας ε, στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Γιατί δεν θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να υποβάλλετε υποψηφιότητα για το Βουλγαρικό Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν έχετε την 15η πείρα. Μπορείτε όμως να υποβάλλετε την ε, υποψηφιότητα για το Ελεκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι έχετε αυτά τα προσόντα. Επίσης, μετά την ε, τριετή κατάρτιση που είχατε στο Πανεπιστήμιο, περάσατε σε ένα από τα πιο σημαντικά, ένα από τα τρία πιο σημαντικά σχέδια στο, Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων. Είπατε ότι στο Υπουργείο αυτό, μετά από τρία μόνο χρόνια κατάρτισης, αναλάβατε στο Βουλγαρικό Γεωργείο Υπουργές μια σειρά εξπός τελέχου. Μιλήσατε για συντονισμό, για αξιολόγηση αποτελεσμάτων, για παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πιο λεπτομεριακά το ρόλο σας στο πολύ αυτό σημαντικό σχέδιο στο Υπουργείο Γεωργίας που μάλιστα αναλάβατε μετά από ελάχιστη φίτηση στο Πανεπιστήμιο, μετά από τριετή από ό,τι βλέπω. Σε ό,τι αφορά την το διορισμό σα ενώ ήσασταν αντιπρόεδρο τη ε, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Μετά από την εμπειρία σα και τα ντοσιά που παρακολουθήσατε, μπορείτε να μα δώσετε ένα είδου χρονική πρόβλεψη. Φυσικά είναι εντυπωσιακό το βιογραφικό σας, ε, αλλά ε, γιατί τώρα που είσαστε στην Κοκομπού υποβάλατε την υποψηφιότητα για ηλεκτρικό συνέδριο. Δεν σας ενδιαφέρει πια η κοκομπού. Επίσης, βλέπω ότι είχατε σημαντική πολιτική θέση. Είπατε ότι θα παραιτηθείτε από οποιαδήποτε πολιτική θέση εφόσον επιβεβαιωθεί ο διορισμό σα. γιατί η συνθήκη της Λισαβόνα απαιτεί ανεξαρτησία για όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Εσεί, έχετε και λόγω του νεαρού της ηλικίας σας κάπως περιορισμένη πολιτική πείρα. Φαντάζομαι ανοίγεται μπροστά σα ένα λαμπρό πολιτικό μέλλον. Μήπως όμως αυτό δημιουργήσει κάποιες πιέσεις ε, πάνω σας εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης ή εκ μέρους άλλων φορέων ή οργανώσεων. Πώς ε, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να ασκήσετε πλήρως την υποχρέωση αυτή ανεξαρτησίας ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης, ε, στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων αναφέρονται δύο επιχειρήσεις. Η Ericsson, φαντάζομαι παραιτηθήκατε από εκεί, όταν εκλέγει, εκλέγει κάτι αλλά αναφέρεται και, μία, και ένα βουλγαρικό μεσητικό γραφείο. Και βλέπω ότι ε, ασχολούσαν με αξιολόγηση, διαχείριση κινδύνων για υπόθηκα δάνεια, συμβάσεις. Τι, ποια είναι η σχέση σας με αυτό το βουλγαρικό μεσητικό γραφείο, γιατί δεν αναφέρεται αυτό στην επαγγελματική σας πείρα. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Ιβάνοβα για να απαντήσει. Uh, Ευχαριστώ. Θα απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν οι ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη χρονική διάρκεια της επαγγελματικής μου εμπειρίας. Πράγματι δεν έχω 30 χρόνια εμπειρίας. Αν είχα 30 χρόνια εμπειρίας θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να είχα ξεκινήσει περίπου 7 ετών να εργάζομαι κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις ε, νομικές απαιτήσεις στην Ένωση. Και σοβαρά τώρα, ε, δεν νομίζω ότι πουθενά στη συνθήκη να αναφέρεται απέτηση για συγκεκριμένη διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας που πρέπει να διαθέτει υποψήφιος. Εάν υπήρχε τέτοια απέτηση, δεν θα είχα κάνει κανέτηση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να βλέπουν έναν υποψήφιο όχι μόνο από την οπτική γωνία της διάρκειας ε, της εμπειρίας, δηλαδή όχι μόνο ποσοτικά, να βλέπουμε την εμπειρία του, αλλά και ποιοτικά και πιστεύω ότι η ποιότητα των 12 αυτών ετών είναι αρκετά υψηλή, ούτως ώστε να καλύψει τις απαιτήσει που υπάρχουν για ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και θεωρώ ότι λόγω της ποικιλομορφής εμπειρίας είναι καλή εμπειρία και θα σας έλεγα κυρία Συγήτρια ότι είπατε επανειλημμένα ότι η ποικιλομορφία είναι πολύ σημαντική κυρίως ε, όταν αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και έχω αυτή την ποικιλομορφία και την, στην εμπειρία όχι μόνο στον κυβερνητικό, στον έλεγχο στο δημόσιο τομέα και στον ειδικό τομέα. Ε, κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα καλό και έχω και εμπειρία και σε αυτή την ε, επιτροπή. Οπότε η απάντησή μου όσον αφορά τα 12 χρόνια είναι αυτή. 12 ποιοτικά χρόνια εμπειρίας που θεωρώ ότι ταιριάζουν στο ρόλο και τη θέση ενός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου. Τώρα όσον αφορά το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν είμαι σίγουρη αν κατανόησα πλήρως την αναφορά που κάνατε όσον αφορά το τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Πήρα το πτυχίο μου κανονικά από το Πανεπιστήμιο, πέντε χρόνια για το πτυχίο, ένα μάστερ, πρώτα πήρα το μπάτσελορ, μετά πήρα το μάστερ όσον αφορά τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, μετά είχα διάφορες άλλες θέσεις μαθητείας που δεν θεωρούσα ότι έπρεπε να αναφέρω, είχα και άλλη εμπειρία πριν εργαστώ στο Υπουργείο και ο συγκεκριμένος ρόλος που είχα ήταν ακριβώς ο συντονισμός της γενικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων, προετοιμασιών. Είναι πολύ μακρύ πρόγραμμα, δεν κρατά ένα-δύο μήνες, αλλά μερικές εβδομάδες. Είναι ένα πρόγραμμα που κρατά χρόνια. Και η γενική προετοιμασία και οι διαπραγματεύσεις ήταν αυτές. Δηλαδή έπρεπε να συντονίζω όλα τα τμήματα του Υπουργείου που σχετιζόταν με τους διαφόρους τομείς που συζητούνται. Τομείς όπως ε, αγορά, κτήματα, αξία των γεών του χρηματορίου, ε, άρδευση, δασοκομεία, επιδοτήσεις κρατικές της γεωργίας, χρηματοδότηση της υπαίθρου, διάφοροι τομείς ε, του αγροτικού τομέα, υπέκυντος σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις και ο ρόλος μου ήταν σημαντικός, διότι έπρεπε να κατανοώ κάθε πρόβλημα, κάθε τομέα και να μπορώ να τα μεταφράσω τα προβλήματα και να τα συνοψίζω για να, να ετοιμάζω τον Υπουργό, τα ανώτερα στελέχη και να ετοιμάζω την ομάδα του Υπουργείου για τις ε, διαπραγματεύσεις. Ήταν σημαντικό έργο διότι όπως προανέφερα θα έλεγα ότι έβαζε τα θεμέλια ούτως ώστε να ετοιμαστεί όλος το τομέας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι πολλές μεταρρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν και αυτή η συνεχής δουλειά με έμαθε πολλά. Όχι μόνο τεχνικά πράγματα, αλλά με έμαθε να συνεργάζομαι με ανθρώπους, ε, να δημιουργώ ομάδες, να εργάζομαι σε ομάδες, που θεωρώ ότι είναι κάτι που ε, σχετίζεται άμεσα με τη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου. Όσον αφορά το ερώτημα κατά πόσο τα ενδιαφέροντά μου για το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού ε, αν υπονομεύθηκε διότι ήθελα να, ε, προ, προκλήθηκε ήθελα να είμαι μέλος, όχι, διότι ξεκίνησα σταδιακά, ξεκίνησα ως κοιόδηση συγγήτρια για κάποιες εκθέσεις. Ε, συνεργάστηκα επικοδομητικά με πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής από πολλές πολιτικές ομάδες και λέω με κάθε πεποίθηση ότι πάντα μέσω συνεργασίας και για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, καλύτερης δυνατής εκθέσεως, μέσω των εργασιών της Επιτροπής, κατέβαζε τέτοιε προσπάθειε. Συνεργάστηκα με άλλε επιτροπέ τη εσωτερική αγορά, προστασία του καταναλωτού, γνωμοδοτήσει για τρόφιμα για τα βρέφη κλπ. ΦΠΑ, διάφορα άλλα θέματα που δεν σχετίζονται με τα θέματα ελέγχου του προπολογισμού. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι είχα κάποιο ενδιαφέρον, ε, είχα κάποια συμφέροντα μέχρι κάποια ημερομηνία και γι' αυτό ξεκίνησα να δουλεύω ενδιαφερόμουν πρωταρχικά για αυτή την επιτροπή και θα εξακολουθεί να με ενδιαφέρει όσο είμαι εδώ. Όσον αφορά τις θέματα των ε, πολιτικών θέσεων, όχι δεν έχω ανώτερη θέση πολιτική και απάντησα έτσι διότι αν απαιτηθεί να παρετηθώ ή να αναστείλω την συμμετοχή μου, να πάψω να είμαι μέλος, θα το κάνω, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είμαι εντελώ ανεξάρτητη. Δεν έχω συζητήσεις και επαφές που σχετίζονται με την πολιτική μου θέση. Σχέσεις που να έπρεπε να αναφέρονται στην αίτηση. Εάν απαιτηθεί, το επαναλαμβάνω, θα σταματήσω να είμαι μέλος, αλλά είναι μια απλή συμμετοχή με ένα απλό μέλος και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν και τώρα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που διατήρησαν τη θέση τους και είναι μέλη κάποιων πολιτικών δομών. Όσον αφορά λοιπόν την ανεξαρτησία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσον αφορά την εταιρεία που αναφέρατε, δεν είμαι σίγουρη ποια αναφέρατε. Θα μπορούσατε να το ξεκαθαρίσετε, να μου πείτε ποιο όνομα αναφέρατε. Γιατί εργάστηκα για διάφορε εταιρείε. Είχα την καλοσύνη να μου πείτε. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Αν διαβάζω καλά, όχι καπροπόρτουκ. Δεν ξέρω, δεν είμαι κανεί να διαβάσω το κυριλικό αλφάβητο. Όχι ποπόρτουκ Μήπως Ντέσα πρόπερτης. Α, Ντέσα πρόπερτης. Ήτανε προσωρινή θέση εκεί που δεν την ανέφερα πουθενά. Ε, ήτανε μόνο για μερικούς μήνες. Και ήμουνα και έγκυος στο πρώτο μου παιδί ε, και δεν θεωρούσα ότι ήταν απαραίτητο να το αναφέρω και να το συζητήσω. Ουδέμια σχέση έχει με το παρόν θέμα. Äh, Σας ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα για την απάντηση των ε, ερωτήσεων αυτών. Η κυρία Γκρέσλε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ότι κυρία συνάδελφε, χαιρόμαστε όταν ε, κάποιος από εμά έχει την ε, ευκαιρία να πάει στο ελεγκτικό συνεδρίο, ειδικά όταν είναι γυναίκα, καθώς έχουμε μόνο δύο γυναίκες και 25 άντρες. Και Ταυτόχρονα είναι και τα νεότερα μέλη οι δύο γυναίκες, ε, η κυρία Καγιουλάιτη ήταν 34 ε, ε, ετών, ούτε και αυτή είχε 15 χρόνια εμπειρία. Και ο κύριος Δέος ο Ιρλανδός συνάδελφος ήταν 33 ετών εκείνος νομίζω, οπότε ακούμε ένα επιχείρημα το οποίο δεν είχε ακουστεί ποτέ σε καμία άλλη ακρόαση, εγώ δεν το είχα ξανακούσει ως θέμα. Και από και όλες. Θεωρώ πως έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μία καλή ε, υποψήφια. Εγώ θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά την άποψή σας για το ελεκτικό συνέδριο. Τι θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει, είπατε πως θέλετε να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο, βεβαίως ε, αλλά πείτε μας λίγα περισσότερα. Και το δεύτερο αφορά την Βουλγαρία, ένα από τα νεότερα κράτη-μέλη ε, που έχει μεγάλα προβλήματα και άρα είναι σημαντικό για εμάς να μάθουμε ποιον ρόλο βλέπετε εσείς ότι μπορείτε να παίξετε όσον αφορά την ε, Βουλγαρία. Υπήρχε και μια δική σας μελέτη για τα προβλήματα των νέων κρατών μελών, οπότε θα ήθελα να μας πείτε πώς ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να προωθήσετε την επαφή του ελεγκτικού συνεδρίου με τη Βουλγαρία. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλε. Αναφερθήκατε στο νεαρό της ηλικία. Να σας υπενθυμίσω πως ο πρώτος ε, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Τέοντορ Χόις, ε, είχε πει πως η νεότητα είναι η μόνη ασθένεια η οποία μέρα με τη μέρα καλυτερεύει. Οπότε, Ακούσατε τις ε, ερωτήσεις ε, της κυρίας Γκρέσλε. Κυρία Ιβάνοβα, παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση για το όραμά μου για το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να χωρίσω την απάντησή μου σε δύο τμήματα. Καταρχήν πιστεύω ότι μέσα στα χρόνια λειτουργίας του το ελεκτικό συνέδριο πέρασε από μια μεταρρυθμιστική διαδικασία της ε, αυτοαξιολόγησης και του peer review της ε, αξιολόγησης ομοτήμων και μετά ε, από τα έγγραφα που διάβασα και από τις συστάσεις ε, που μελέτησα διαμόρφωσα και τη δική μου γνώμη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ελεκτικό συνέδριο να συνεχίσει και να βαθύνει την επικοινωνία του με τα βασικά στελέχη της, της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή για να καταλάβει τις ανάγκες τους και να μπορέσει να τις ε, αντιμετωπίσει και να τις ικανοποιήσει. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση οδεύει το ελεκτικό συνέδριο και θα πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης ε, έγιναν πολλές εκκλήσεις και από την Επιτροπή αυτή και στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης και του peer review ε, εκκλήσεις για ε, ενημέρωση των διαφόρων εκθέσεων, για απόσπαση των διαφόρων εργαζομένων, να μην μένουν πολλά χρόνια στην ίδια θέση, να υπάρχει μια μετακίνηση και νομίζω ότι και το ελεκτικό συνέδριο προ αυτή την κατεύθυνση κινείται. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ενισχυθεί. Δηλαδή το ελεκτικό συνέδριο να δώσει μια συνέχεια στις συστάσει που εκδίδει, δηλαδή να μην εκδίδει μια σύσταση και μετά να την ξεχνά. Θα πρέπει να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει πρόοδος και από αυτή την άποψη στο ελεκτικό συνέδριο και τέλος, εξίσου σημαντικό όμως θέμα, είναι οι δείκτες επιδόσεων, οι δείκτες απόδοση. Από ό,τι ξέρω, το ελεκτικό συνέδριο προτίθεται να σημειώσει πρόοδο και στην κατεύθυνση αυτή, να ενισχύσει δηλαδή τους μηχανισμούς που προσδιορίζουν το σημαντικό ρόλο των δικτών αυτών επιδόσεων. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα της προσωπικής μου απόψης και το προσωπικό μου όραμα για το ελεκτικό συνέδριο, Νομίζω ότι πέρυσι, την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για το ποια άγουσα θα πρέπει να ακολουθήσει το ελεκτικό συνέδριο. Σίγουρα ο έλεγχος απόδοσης θα πρέπει να αποκτήσει όλο και μεγαλύτερο ρόλο και θα δώσω μάχη για να καθιερωθεί κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα για τι ειδικέ εκθέσει. Το είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια. Θα ήθελα να δίνονται πιο έγκυρα, να είναι πιο ελαστικέ, να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και να ε, καταλήγουν σε πιο συγκεκριμένες συστάσεις, όχι μόνο σε γενικές και όρισες δηλώσεις ότι κάτι πάει στραβά, να προκύπτουν συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νομίζω ότι εκεί έγκυται η ιδιαίτερη αξία μιας ειδική έκθεσης. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε το όλο και μεγαλύτερο και ενισχυμένο ρόλο των χρηματοδοτικών μηχανισμών, των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών και αναφέρθηκε και από το ελεγκτικό συνέδριο η πρόθεση να διενεργηθούν έλεγχοι και προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιος είναι ο ρόλος των νέων μακροχρηματοπιστωτικών ε, οργάνων και εργαλείων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δημόσια κρόση που οργανώσαμε και πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον που προκάλεσε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για αυτό γιατί όντως το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε 110 δισεκατομμύρια ε, ευρώ υποχρεώσεις για τον κοινωτικό προϋπολογισμό από το ισοζύγιο πληρωμών και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και τα κονδύλια αυτά, μπορώ να το πω και ε, δημοσίως, ε, τα ποσά αυτά δεν ελέγχονται σωστά. Δεν ελέγχονται με αρκετή διαφάνεια. Δεν υπάρχει αρκετό δημόσιο έλεγχο. Πιστεύω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και το Ελεκτικό Συνέδριο να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτόν τον έλεγχο. Γιατί μιλούμε για ε, κοινοτικά κονδύλια. Θα πρέπει να ελέγχεται η διάθεσή του. Ό,τι αφορά τι αιτήσει απαλλαγέ και τη δήλωση αξιοπιστία, τον ΤΑΣ. Πολλέ φορέ τα μέλη τη Επιτροπή και εγώ ίδια απευθύναμε έκκληση στο ελεκτικό συνέδριο να μας δίνει σαφέστερη ανάλυση για, για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών. Βέβαια, συνειδητοποιώ ότι δεν είναι εύκολο αυτό το έργο και απαιτούνται πολλοί πόροι. Είναι πολύ δύσκολο να διεκπαιρεωθεί, αλλά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να δίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφείς αναλύσεις για, προβληματικά, για προβληματικούς τομείς στο Ευρω... στο... στα διάφορα κράτη-μέλη, για το είδος των λαθών που πραγματοποιούνται από τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβούν σε σαφή ανάλυση εμπεριστατωμένη. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πτυχές, θα ήθελα να αναφέρω τη σχέση με τους εθνικούς φορείς ελέγχου και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς φορείς ελέγχου, Νομίζω ότι και από τη διακήρυξη της Λίμα ζητήθηκε εντατικοποίηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ε, φορέων ελέγχου και του ελεκτικού συνεδρίου. Και ένα καλό παράδειγμα ήταν η ακρόση που είχαμε για το Μηχανισμό Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτική Σταθεροποίηση, ESM και ESFM. Είχαμε εκπροσώπου από το Γερμανικό και από το Ολλανδικό Ελεκτικό Συνέδριο. Και αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Τέτοιου είδου ανταλλαγέ είναι πραγματικά ανεκτήμητε και θα τι προωθήσω ιδιαίτερα να εκλεγώ, αν επιβεβαιωθεί ο διορισμό αν επιβεβαιωθεί ο διορισμό μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να υπολογίσετε πάνω μου, μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη ότι θα ασχοληθώ και θα, θα προσπαθήσω να βελτιωθούν αυτέ οι σχέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα στη διάρκεια τη δημόσια ακρόαση, ρώτησα τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Καλντέιρα, και θα το ε, επαναφέρω αυτό το ζήτημα αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου. Δεν μπορούμε να οργανώνουμε πιο τακτικά ανταλλαγές απόψεων, κοινέ συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και των εκπροσώπων του Ελεκτικού Συνεδρίου. Νομίζω ότι μπορούν να γίνονται και οι ειδικέ τέτοιε συσκέψει για επιμέρου θέματα. Γιατί σε τέτοιου είδου ανταλλαγέ απόψεων μπορούν να προκύψουν ιδέε και να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκε των μελών τη Επιτροπή. Αυτές λοιπόν είναι οι σκέψεις μου και το όραμά μου ε, για τις μελλοντικές προκλήσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση για τη Βουλγαρία, νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχω αποδείξει και θα συνεχίσω να το κάνω ότι είμαι ουδέτερη άσχετα από το που λαμβάνει η χώρα ένα σφάλμα, ένα σφάλμα είναι σφάλμα και θα πρέπει να εντοπίζεται και να καταγράφεται, άσχετα με το ποια χώρα το διαπράττει. Φυσικά, ο διάλογος και η επικοινωνία είναι σημαντική μεταξύ των εθνικών ελεκτικών φορέων και θεσμών και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Όπως είπατε, κυρία Γκρέσλερ, ήμουν εισηγήτρια για τη μελέτη σε ό,τι αφορά τα πρωτεξιακά κονδύλια για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Μπορεί η Επιτροπή να μην το ξέρει, αλλά προσκάλεσα και τον συνάδελφο Φιέλνερ στη Βουλγαρία στη διάρκεια της ε, φετινής διαδικασίας απαλλαγής για να γίνει διάλογος και με τις αρμόδιες αρχές και να αντιληφθούμε πού έγινε τα προβλήματα, πού έχει σημειωθεί πρόοδος, γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα που τον δέχτηκε παρά τις προσπάθειες ε, που έγιναν για τη διαδικασία απαλλαγής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να παρακαλέσω τώρα για να προγραμματίσουμε να μου πείτε ποιοι θέλουν το λόγο. Μιούλτερ, ο Τζι, Κάλβιν και η παράκλησή μου είναι στις ε, απαντήσεις να είμαστε και λίγο πιο σύντομοι για να μείνουμε εντό του προγράμματος. Κύριε Μιούλτερ, ευχαριστώ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση για την ε, συναδελφό την κυρία Ιβάνοβα. Μία από τις πιο προβεβλημένες εκθέσεις ε, του Ελληνικού Συνεδρίου είναι η ετήσια έκθεση όπου βεβαίως υπάρχει μια γνωμοδότηση για το αν πρέπει να δοθεί ε, θετική ή αρνητική δήλωση εξοπιστίας και είναι λυπηρό το ότι τα τελευταία 17 χρόνια ήταν αρνητική αυτή η δήλωση. Εάν ε, μπορούσε να κάνει η κυρία Βάνοβα ότι ήθελε τι θα ε, συνιστούσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε θετική δήλωση εξοπιστίας. Πολύ απλή ερώτηση. Ευχαριστούμε κύριε Μίλντερ. Ε, παρακαλώ απαντήστε σύντομα. Ευχαριστώ. Είναι σύντομη αλλά δεν είναι εύκολη ερώτηση, είναι πολύ σοβαρή είναι μία από τις σοβαρότερες ε, ερωτήσεις που προσπαθούσαμε να απαντήσουμε στην Επιτροπή αυτή και νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι μόνο ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα που καταβάλουν προσπάθειες και ζητούμε συνεχώς να γίνονται εθνικέ δηλώσει, διαχείριση. μεγαλύτερη ευθύνη από πλευρά κρατών μελών. Δυστυχώ, φέτο, είδαμε εκ νέου ότι κανένα κράτο μέλο, εκτό από τη Βουλγαρία δεν ήθελε καν να μιλήσει με τον εισηγητή. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η τάση. Εξαρτάται όμω κατά πολύ από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εξακολουθεί να πιέζει προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει η συζήτηση όσον αφορά την ηλικία, διότι, κύριε Πρόεδρε, κάνατε σωστή σκέψη. Και εμείς λέμε ότι η νεολαία δεν είναι θέμα ηλικία, η νεότητα δεν είναι θέμα ηλικία Και είμαι ευτυχή για την υποψηφιότητα τη κυρία Ιβάνοβα. Θεωρώ ότι έχει μια προσωπικότητα άκρως ενδιαφέρουσα. Έχει εμπειρία μεγάλη και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και χαίρομαι που η κυβέρνησή της την πρότεινε. Έχει τις ε, γνώσεις, τις ικανότητες, έχει την εμπειρία. Πράγματι είναι η εμπειρία που δεν είναι 15 ετή, όμως σημαντική εμπειρία και οι εμπειρίες αποκτώνται. Εξελέξαν πρόεδρο της Δημοκρατίας που κατά τη διάρκεια της ε, ε, εκστρατείας είπαμε ότι δεν έχει υπουργική εμπειρία. Εξελέγει όμως. Η εμπειρία είναι σημαντικό αλλά δεν είναι τα πάντα. Έχετε παρόλα αυτά πολύ καλή εμπειρία. Έχετε την ανεξαρτησία Μιλήσαμε ότι ανήκετε, για το ότι νίκετε σε ένα πολιτικό κόμμα. Εγώ δεν έχω συμβουλή να δώσω, αλλά θεωρώ ότι για ένα μέλος του ελεκτικού συνεδρίου που έχει καθήκοντα σημαντικότατα για μας, κάθε, πώς να το πω, κάθε συμμετοχή, κάθε σύνδεση που θα μπορούσε ακόμα και εικονικά ε, να δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν είναι κανείς ανεξάρτητος, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει, διότι χρειαζόμαστε μέλη που είναι πραγματικά ανεξάρτητα. Θα ήθελα να σταματήσω αφορά το θάρρο. Εμεί χρειαζόμαστε ένα ελεκτικό συνέδριο γενναίο, θαραλέο. Το ερώτημά μου αφορά την απαλλαγή και τον έλεγχο του Συμβουλίου. Δεν ξέρω ποια καθήκοντα ανατεθούν εντό του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά εκπλήσωμαι διότι σε συζητήσει που κάνουμε βλέπω ότι υπάρχει απόκληση ότι κατηγορεί για πολλά το Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου Προβλησμού και δεν κάνει πολλά πράγματα το ελεκτικό συνέδριο τελικά. Αν επιφορτιστείτε με τους ελέγχους ή αν γνωμοδοτείτε σαν μέρος του σώματος, σαν μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, πώς θα εκφράσετε τις απόψεις σας όσον αφορά την απαλλαγή προς το Συμβούλιο, θα έχετε αυτό το θάρρος, αυτή τη γενναιότητα δεν θα έλεγα ότι δεν είναι γενναίο το ελεκτικό συνέδριο, αλλά εκπλήσωμαι από τα λίγα πράγματα, τις λίγες καταγγελίες που κάνει απέναντι στο Συμβούλιο. Θα έχετε αυτό το θάρρος. Ούτω ώστε το ελεκτικό συνέδριο να το τραβήξετε προς μια αξιολόγηση πολύ ανεξάρτητη, όταν κάτι δεν πάει καλά να το λέει και να αλλάζουν τα πράγματα, αν δεν πηγαίνουν καλά. Ευχαριστούμε κύριε Οντή. Κύριε Ιβάνοβα, παρακαλώ, απαντήστε και σε αυτές τις δύο ερωτήσεις σύντομα. Ναι. Κύριε Ντί, μπορείτε να βασιστείτε πάνω μου. Είμαι, όπως είμαι και σε αυτή την Επιτροπή, είμαι αντικειμενική και ουδέτερη. Θα συνεχίσω να είμαι το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ένα σφάλμα είναι ένα σφάλμα, τα σταλία είναι τα σταλία ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία συμβαίνει, το θεσμικό όργανο στο οποίο συμβαίνει. Νομίζω ότι ο ρόλο ενό μέλου ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου είναι να εντοπίζει το σφάλμα και να μην ε, φοβάται, να μην υποκρίνεται σαν να μην έχει συμβεί κάτι. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μου λοιπόν. Ε, το ίδιο θα κάνω αν εκλεγώ ω μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Σα ευχαριστώ για τη σύντομη απάντηση. Κάλβιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ιβάνοβα για την υποψηφιότητα. Είχα την χαρά να συνεργαστώ μαζί της στην Επιτροπή μας τα τελευταία τρία χρόνια. Για λόγους ε, συνέπειας βεβαίως θα θέσω το ίδιο ερώτημα το οποίο θέτω κάθε φορά και αφορά την ερμηνεία της συνθήκης της ε, Λισαβόνας λέγεται πως θα πρέπει, αναφέρει η συνθήκη πως θα πρέπει να έχουν τα ειδικά προσόντα για το αξίωμά τους τα α, μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και το ερώτημά μου είναι πώς το ερμηνεύετε. ποια είναι αυτά τα ειδικά προσόντα. Κατόπιν, ποιες ήταν οι διευθυντικές θέσεις που κατήχατε και τρίτον, αναφέρατε πάρα πολλές φορές τον έλεγχο απόδοσης και αυτό είναι σημαντικό γιατί στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου μιλάμε για την απόδοση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συγγραφτές απαντήσεις ε, ε, δώσατε βεβαίως ε, έναν ορισμό του έλεγχου απόδοσης, ο οποίος όμως δεν είναι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή το ελεγκτικό συνέδριο. Ποιες είναι οι αλλαγές που θεωρείτε πως πρέπει να γίνουν για να αρχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριε Κάλβιν κυρία Ιβάνοβα. Αν θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Απαντήστε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα για τα ιδιαίτερα αυτά προσφόντα. Νομίζω πως ε, είχαμε μια καλή συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για την εντολή των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου και με ικανοποίησε ιδιαίτερα η απάντηση της κυρίας Πετροσκεβιτσιένη, η οποία είπε πως ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να γνωρίζει τον έλεγχο, να τον αντιλαμβάνεται, να έχει δουλέψει πάνω στο αντικείμενο και να συνεργάζεται στο πλαίσιο μια ομάδα. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα σώμα 27 μελών, θα πρέπει να μπορεί κανείς να εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας και να προωθεί τις ιδέες του, να τι υπερασπίζεται, αλλά ταυτόχρονα να είναι ευέλικτο, ε, να μπορεί να συμβιβαστεί για να επιτύχει τους ε, στόχους ε, και να καταλήγουμε τελικά σε μια απόφαση. Εγώ δεν θεωρώ πως ε, έχω αυτά τα προσόντα. Θα πάω και λίγο παραπέρα από αυτά τα οποία λέμε συνήθως για τις τεχνικές απαιτήσεις. Νομίζω πως είναι σημαντικό Εντάξει, οπωσδήποτε η έλεγχη, η χρηματοοικονομική και η έλεγχη συμμόρφωση, αλλά και η έλεγχη της ε, απόδοσης, όπως αναφέρατε, είναι κάτι το αναγκαίο για να είναι πλήρης ο έλεγχος και νομίζω πως προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και να εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ποια είναι, πού πάνε τα λεφτά του. Όλα αυτά τα λεφτά που ξοδεύονται, ξοδεύονται σωστά, αλλά και με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό. Και ακριβώς αυτός είναι ο ορισμός ο οποίος έχω δώσει για τον έλεγχο, για την αποτελεσματικότητα και την ορθή χρήση αυτών των κονδυλίων. Δεν είναι όπως είπε η κυρία Γιάλα ακριβώς να ξοδέψουμε κάποια λεφτά, αλλά να πάνε σε έναν σωστό σκοπό για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών σε τελική ανάλυση. Αυτό είναι νομίζω ο τελικός στόχος. Τώρα για διευθυντικέ θέσει. Διευθυντή συγκεκριμένα δηλαδή δεν ήμουν ε, κάπου με αυτό τον τίτλο, αλλά έχω διευθύνει ομάδες και τι έχω οργανώσει κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε και με καλά αποτελέσματα. Για τον έλεγχο δε της ε, απόδοσης νομίζω πως ήδη απάντησα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Ιβάνοβα για την απάντηση των ερωτήσεων του κυρίου Κάλβιν. Τώρα, εάν ε, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τότε... Κλει... Α, με συγχωρείτε κύριε Γκάιερ. Ναι, μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση γιατί περίμενα να το πει κάποιος συνάδελφος αλλά δεν το είπε. Είδα το βιογραφικό σας κυρία Ιβάνοβα και διαπίστωσα πως σε τρία χρόνια είχατε πέντε διαφορετικές θέσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσετε εσείς ε, πώς εξηγείται αυτή η γρήγορη αλληλουχία ε, θέσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάιρη. Κύριε Ιβάνοβα. Αν αναφέρεστε στις θέσεις μου στι Ηνωμένε Πολιτείε σε διάφορε επιχειρήσεις, ναι, στη ΣΥΠΑ είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στην Ευρώπη. Και για οικονομικούς λόγους χρειάστηκε να μετακομίσω από μια πολιτεία σε άλλη, μερικές φορές λόγω του συμβολέου που είχα αυτό είναι ο λόγο. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Τώρα, ε, υπάρχει κάποιος άλλος ε, συνάδελφος πριν την εισηγήτρια. Όχι, οπότε η κυρία Νίσα Γιαλασέντερ έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για όλες τις απαντήσεις που έδωσε και θα ήθελα να πω ότι πέραν των ουσιαστικών θεμάτων που έθιξε και μάλιστα μερικά περιλαμβανόταν και στις απαντήσεις που έδωσε για γραπτός, μερικά αφορούσαν και τα οργανωτικά. Γιατί ξέρετε στις συζητήσεις που έχουμε με το ελεκτικό συνέδριο Θέλουμε περισσότερη παρουσία προσωπικού. Βέβαια όλα τα θεσμικά όργανα έχουν ε, έλλειψη προσωπικού και το ελεκτικό συνέδριο το ίδιο. Θα θέλαμε περισσότερο προσωπικό να αφιερώνεται σε τέτοια καθήκοντα επιχειρησιακού ελέγχου. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη να σας θέτουμε τέτοια ζητήματα, γιατί δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι θα γίνετε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά πιστεύετε ότι ε, μπορείτε να μειώσετε το δικό σας γραφείο ώστε να απελευθερωθούν ε, ανθρώπινοι πόροι για το επιχειρησιακό σκέλος. Έχετε μια τέτοια πρόθεση και σε περίπτωση που διοριστείτε, σε ποια ομάδα του ελεκτικού συνεδρίου πιστεύετε ότι θα αξιοποιήσετε καλύτερα την εμπειρία σας. Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες, σε ποιο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου πιστεύετε θα υπηρετήσετε καλύτερα. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Κύριε Ιβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αγιάλα, για την πρώτη ερώτηση. Ναι, θεωρώ πως το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει βεβαίως να δίνει το καλό παράδειγμα ε, όσον αφορά αυτά τα οποία απαιτεί από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους πολίτες. Γίνονται περικοπές και πρέπει να γίνουν και στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο δεύτερο ερώτημα που θεωρώ ότι μπορώ να καλύτερα Προσπάθησα να εξηγήσω πως δεδομένης της πείρας μου θεωρώ πως μπορώ να προσφέρω ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μυστήριο καμιά φορά για κάποια μέλη της Επιτροπής αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης τα χρηματοπιστωτικά μέσα για μακροοικονομική βοήθεια, δεδομένης της πείρα μου σε ελέγχου ε, απόδοση και εκεί πέρα νομίζω πως μπορώ να προσφέρω και μπορώ να σα υποσχεθώ πως θα, θα προσπαθήσω να γίνουν πιο γρήγοροι αυτοί οι έλεγχοι και βεβαίω ε, να ανταποκρίνονται περισσότερο και σε αυτά τα οποία θέλουν τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα που απαντήσατε και αυτές τις ερωτήσεις. Ε, τελειώνει εδώ πέρα το τμήμα της δημόσιας ε, συζήτησης. Θα περάσουμε στην αξιολόγηση που θα είναι και των θυρών. Γι' αυτό σας παρακαλώ ε, όλοι όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής και δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα για τις απαντήσεις που έδωσε. Σας ευχαριστώ πολύ.